Το λόγο έχει η κυρία Συγκήτρια. Παρακαλώ κυρία Πακ. So. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πακ, νομίζω ότι μπορώ να αρχίζω σιγά σιγά, έτσι, πάμε. Αγαπητή κυρία Επίτροπε, αγαπητέ Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, αγαπητοί παρόντες ακόμα συνάδελφοι, φεύγουν και οι νέοι μας, κρίμα, γιατί ε, ε, μιλάω για κάτι που θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο στόχος ή στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για αύξηση της απασχολησιμότητας δεν πρόκειται να επιτευχθούν χωρίς την παιδεία, και την επίσημη αλλά και την άτυπη ε, μόρφωση. Και είμαι βέβαιη και χαίρομαι που και τα τρία θεσμικά όργανα επιφυλάσσουν στην παιδεία το ρόλο που τις αναλογεί και συμφώνησαν να αυξηθεί κατά 40% ο προϋπολογισμός, η γλωσσομάθεια, η εκμάθηση ξενογλωσσών η απόκτηση ε, προσόντων και δεξιοτήτων είναι πάρα πολύ πολύτιμα σήμερα, ιδιαίτερα για τους ε, νέους της Νότιας Ευρώπης που δεν έχουν ε, εργασία. Θα μπορούσαν να βρουν δουλειά σε άλλη χώρα εάν γνωρίζανε μια ξένη γλώσσα και είχαν δεξιότητες συμβατές με την πολυπολιτισμικότητα. Το πρόγραμμα στην πρότασή του είχε ένα τίτλο που δεν μπορούσα ε, να το καταλάβω. Τι θα πει Εράσμους για όλους. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υφίσταται. Γι' αυτό χαίρομαι που τελικά από κοινού καταφέραμε να βρούμε ένα τίτλο που να περιγράφει ε, και να καθιστά κατανοητό αυτό το πρόγραμμα. Έρασμος ΣΥΝ. Δεν είχε ενθουσιαστεί ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο, αλλά τελικά νομίζω ότι συμφωνήσαμε. Να σας πω κατά τη διάρκεια της συζήτησης τι ήταν σημαντικό για μας. Ακούσαμε τους νέους μας που ε, συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα, μας είπαν τις αγωνίες τους και τις επιθυμίες τους. Παράδειγμα, είναι πολύ μεγάλη η απήχηση αυτού του προγραμμάτος, του εφόρου προγραμμάτων. Είναι ε, ως ένα σήμα που γνωρίζουν οι πάντες, Κομένιους, Γκρούντ, Λεωνάρδο, ε, συνεχίζουν να ισχύουν τα ονόματα αυτά και πολλά άλλα. Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αρχικά ελάχιστο υπολογισμό και χαίρομαι που έχει αυξηθεί η πυρικοδότηση πλέον για να γνωρίζει κάθε πρόγραμμα τι κονδύλια έχει για το επόμενο διάστημα ε, των 7 ετών και υπάρχει μια ασφάλεια σχεδιασμού και προγραμματισμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, από το 1992 για πρώτη φορά έχουμε το δικαίωμα να συζητάμε καν και να μιλούμε για την νεολαία και για την παιδεία. Μέχρι τότε ε, δεν υπήρχαν ε, αναφορές στη συνθήκη. Γι' αυτό από το 1994 ήρθε το πρόγραμμα Κομμένιος που συνδέει σχολεία μεταξύ τους ε, με την ηλεκτρονική αδελφοποίηση των σχολείων. Ε, μαθητές και δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί μπορούν να εργάζονται στο ίδιο πρόγραμμα. 100.000 νέα σχολεία θα συμμετάσχουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο στην ηλεκτρονική αδελφοποίηση των σχολείων, το e-twinning. Έχουμε λοιπόν ήδη ε, την μεμονωμένη ε, διαδικασία ε, ένας μαθητής από ηλικία 14 ετών και άνω μπορεί να μεταβεί σε μια άλλη χώρα για μια σχολική χρονιά. Λεωνάρδο, είναι επαγγελματική κατάρτιση. Ο αέρασμος διατηρείται και διευρύνεται. Διευρύνεται σε ένα τέτοιο βαθμό που μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Δηλαδή και στα πλαίσια ε, των bachelor και των master και σε διδακτορικό ακόμα, δηλαδή προπτυχιακό, μεταπτυχιακό μέχρι και διδακτορικό. Αλλά είναι πολύ μικρή υποτροφία, 200 ευρώ. Τι να τα κάνεις στο εξωτερικό, ούτε να ζήσεις ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς με 200 ευρώ. Θα πρέπει να υπάρχει και άλλη δυνατότητα λοιπόν και χαίρομαι πάρα πολύ και καλωσορίζω αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυνατότητα δανειοδότησης για να μπορεί κανείς να κάνει όλες τις μεταπτυχιακές του σπουδές σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσφορά είναι αυτό δεν είναι υποχρέωση. Διατηρείται ο έρασμος, αλλά αυτή η προσφορά είναι σημαντική γιατί πολλοί δεν έχουν καν τη δυνατότητα να τα βγάλουν πέρα με αυτά τα 200 ευρώ. Ε, μια τέτοια προσφορά όμως θα μπορούσαν να τη δεχθούν και ως κοινοβούλιο αγωνιστήκαμε και φροντίσαμε να υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια για την αποπληρωμή αυτού του δανείου και ελπίζω πάρα πολύ και εύχομαι να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Βασιλείου, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Ντόρις Πάκ και τους κύριους εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν. Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι πως πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά και αξιοσέβαστα προγράμματα της Ευρώπης. Η οικονομική και κοινωνική κρίση της Ευρώπης έδωσε έκανε ακόμα περισσότερο επίγον την υποστήριξή μας στην εκπαίδευση, κατάρτιση και πολιτική για τους νέους. Και με χαρά μπορώ να πω ότι το κείμενο που συζητούμε σήμερα δικαιώνει τις συλλογικέ μας προσπάθειες. Το 2011 η Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση για ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση κατάρτιση, της νεολαία και τον αθλητισμό υπό το φως της αργής οικονομικής ανάπτυξης, της απαράδεκτα υψηλή ανεργίας των νέων και τεράστιων προκλήσεων που, των τεράστιων προκλήσεων που δημιούργησε η ψηφιακή μετάβαση. Η Επιτροπή με βάση αυτό θεωρούσε ότι το business as usual δεν ήταν επιλογή. Οι δαπάνες μας πρέπει να ταιριάζουν τις πολιτικές προσδοκίες μας. Για να καλύψουμε και αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις μεγάλες προκλήσεις της Ευρώπης σήμερα θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη συμμετοχή των νέων. Αυτό είναι ο λόγος τον οποίο η Επιτροπή είχε προτείνει αύξηση 70% των δαπανών, ε, των υφιστάμενων δαπανών. Ωστόσο είμαι ικανοποιημένη γιατί σε αυτό λάβαμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και τονίζω ότι παρά την συνολική μείωση του προπολογισμού της Ένωσης, ο προπολογισμό για τις πολιτικές αυτές θα είναι 14,7 δις ευρώ την επόμενη επταετία, κάτι που συνιστά αύξηση κατά 40% επί των παρουσών δαπανών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Υπάρχει μια έρευνα για τα προσόντα των ενήλικων στην Ευρώπη και η έρευνα αυτή δείχνει το 20% των, εργαζομε... των ε, ε, ατόμων σε ηλικία εργασίας έχουν χαμηλές ικανότητες ε, αλφαβητισμού και αριθμητικής. Πρέπει να προσφέρουμε νέες δυνατότητες σε αυτούς τους ανθρώπους στο πλαίσιο της τεχνολογίας της πληροφορίας. Σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι. 10% σε κάποιες χώρες, πάνω από 50% σε άλλες χώρες. Ταυτόχρονα και παράδοξα βλέπουμε ότι πάνω από 2 εκατομμύρια κενές θέσει εργασίας στην Ευρώπη ε, μία στις τρεις επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν άτομα με τα σωστά προσόντα. Αυτό είναι ο λόγο τον οποίο χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα προσπαθήσει να βελτιώσει το επίπεδο των προσόντων και ικανοτήτων των ανθρώπων, να εξυγχρονίσει τις δομές μάθησης σε τυπικό και σε άτυπο επίπεδο. Πρέπει να βοηθήσουμε όλους αυτούς να προσφέρουν και να παραδώσουν τα προσόντα που χρειαζόμαστε τώρα και στο εγγύς μέλλον. Το Erasmus Plus προσφέρει μια σειρά καινοτομιών. Πρώτον, στην ανώτερη εκπαίδευση περιλαμβάνει όλα τα περιέχει όλες τις δυνατότητες ε, ε, παροχής βελτίωσης των δυνατοτήτων κάτω από μία δομή. Κάτι που θα ενισχύσει την συνοχή και την ορατότητα της Ένωσης, των δράσεων της Ένωσης και θα κινητοποιήσει συνέργειες. Ταυτόχρονα επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δραστηριότητες για την ε, νεολαία μέσα στο πλαίσιο του building bridges μεταξύ επίσημης και μη και άτυπης εκπαίδευσης. Κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερα στους τομείς αυτούς. Τρίτον, και βάσει και των στόχων μας ενισχύουμε τους δεσμούς μεταξύ της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας κινητοποιώντας νέες εταιρικέ σχέσεις και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην απασχολησιμότητα των νέων. Τέταρτον, για πρώτη φορά για πρώτη πρώτη φορά προσφέρουμε χρηματοδότηση της Ένωσης στον κόσμο του αθλητισμού, βελτιώνοντας τη διακυβέρνησή του για να αντιμετωπίσει απειλές όπως το ρατσισμό, το τοπάρισμα και το στήσιμο παιχνιδιών υποστηρίζοντας, ε, βελτιώνοντας τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πολίτες της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι το νέο πρόγραμμα θα διευρύνει τις ευκαιρίες για τους πολίτες και για την εκπαίδευση στους τομείς αυτούς. Επίσης θα προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες στους φοιτητές και στα πανεπιστήμια και στην επαγγελματική κατάρτιση να περάσουν τμήμα των ε, σπουδών του στο εξωτερικό για να να αποκτήσουν ε, αξιόλογη εμπειρία εργασιακή σε άλλη χώρα. Θα ενισχύσει τις ανταλλαγές νέων και θα ενισχύσει την ε, θελοντική ανταλλαγή νέων σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς και στον τομέα της νεολαίας, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερες ευκαιρίες ενημέρωσης και επικαιροποίησης των προσόντων τους. Το πρόγραμμα θα προσφέρει ευκαιρίες τους, τις οργανώσεις νέων και στα θεσμικά ιδρύματα, να συνεργαστούν με εταίρους σε άλλες χώρες, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να μάθει ο ένας από τον άλλον και να οικοδομήσουν κοινά έργα. Θα προσφέρει υποστήριξη στα κράτη-μέλη για την καινοτομία και, νέες, και νέα ανάπτυξη πολιτικών. Για όλα αυτά πρέπει να αυξήσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των συστημάτων ε, νέων σε όλη την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα έχετε την ευκαιρία να υποστηρίξετε ο, πλήρως ένα νέο φιλόδοξο, φιλόδοξο πρόγραμμα που μπορεί να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων προς το καλύτερο. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ζανίκη, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ε, ε, α, αποουσιάζει Καρβάλιο από την Επιτροπή Προπολογισμών. Μαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επιτροπή. Το να επενδύσουμε στο Εράσμος ισοδυναμεί με επενδύσεις στην νεολαία. Το Εράσμος Plus είναι το νέο πρόγραμμα για την νεολαία ε, και για τον αθλητισμό με στόχο να αυξηθούν οι δεξιότητες ε, και οι γνώσεις των νέων, ε, τονώνοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους. Η ανέργεια των νέων είναι βασικό πρόβλημα σήμερα στην Ευρώπη. Γι' αυτό η Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, εξέτασε κατά προτεραιότητα όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την νεολαία και κυρίως ε, με την απασχόληση των νέων. Το Εράσμους είναι λοιπόν ε, στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο. Τρία δις είναι ο συνολικός περιπολογισμός και η αύξηση ανέρχεται στο 40%. Καταδεικνύεται έτσι η βούληση της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου να επενδύσει στο μέλλον της νεολαίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης, η κυρία Μπλίνκεβιτσούτη, παρακαλώ. Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό πρόγραμμα Erasmus Plus. Είναι αποτέλεσμα που ως εισηγήτρια από την Επιτροπή απασχόλησης ε, είχα θέσει ως στόχο εξ αρχής. Είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό το ότι τώρα υπάρχει καλύτερη δομή του προγράμματος με σαφή υποπρογράμματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικά σε διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επίσης, ξεχωρίσαμε τις ε, δραστηριότητε νέων και τον, ε, τονίζοντας την κατανομή του περιπολισμού, κάτι που αρχικά δεν υπήρχε στο σχέδιο. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση, πέραν της εκπαίδευσης των ενηλίκων. Η επαγγελματική κατάρτιση παίζει όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο στην επίτευξη των στόχων για την Ευρώπη του 2020. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το υψηλό επίπεδο ανεργίας με τον τρόπο αυτό, ενώ θα βοηθήσει και την προώθηση της κουλτούρας, της διαβίου μάθησης για να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και να προωθηθεί η ενεργή λειτουργία του πολίτη. Αυτό απαιτεί βελτίωση συνεχώς των προσωπικών ε, προσόντων και ικανοτήτων. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ εκ νέου ε, το γεγονό ότι πετύχαμε ένα τόσο καλό προγμεράσμος. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματο Επιτροπή Βιομηχανία τώρα η κυρία Τσικάου. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, οι επενδύσεις, οι επενδύσεις στην παιδεία, οι επενδύσεις στην παιδεία είναι βασικό εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκπρόσωπος, ε, ως εισηγήτρια της Επιτροπής ΙΤΡΕ υποστήριξα την πρόταση της Επιτροπής και ζήτησα να εντάξουμε εδώ την βιομηχανική πολιτική της Ένωσης. Η Επιτροπή ΙΤΡΕ ζήτησε να συμπεριληφθούν μεταξύ των στόχων του προγράμματος η κινητικότητα των ατόμων για το ξεκίνημα της επαγγελματικής απασχόλησης, ενώ τονίσαμε τη δυνατότητα επιλεξιμότητας υποψηφίων διδακτόρων σε άλλη χώρα μετέχοντας το πρόγραμμα αυτό είναι σημαντικό να ενισχυθεί η πρόσβαση στα προγράμματα αυτά, στο πρόγραμμα αυτό, ώστε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει νέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση να μπορούν να μετάσχουν. Πρέπει να έχουμε περισσότερα άτομα άνω των 35 ετών που ε, μετέχουν στη διαβίω εκπαίδευση. Είναι σημαντικό τούτο να, να, ορίσουμε σε παράτημα του κανονισμού και όχι σε κατεξοδότηση πράκτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων ακολουθούν ομιλητές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η κυρία Σκουλεύσκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το θέμα που συζητούμε είναι ζωτικό για εκατομμύρια Ευρωπαίων. Σε σύγκριση με το τι είχαμε στο παρελθόν, ο προπολογισμό έχει αυξηθεί. 14 δις στην επταετία. Όλα τα προγράμματα ενσωματώθηκαν σε, κάτω από μία στέγη. Αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην εκταμείευση των πόρων και θα κάνει τις δαπάνες πιο ορθολογικές. Με όλα αυτά ε, τα δεδομένα θα τονίσω ότι η δημιουργία παρότι, μάλλον το γεγονός ότι δημιουργήσαμε ένα νέο πρόγραμμα και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι λύσεις θα πρέπει να ταιριάζουν στους στρατηγικούς μας στόχους. Δηλαδή, τα νέα προγράμματα, οι στόχοι των νέων προγραμμάτων για την εκπαίδευση των νέων πρέπει να επιτρέπουν στους νέους να βελτιώσουν και να καταλάβουν ότι βελτιώνονται οι δυνατότητες απασχόλησής τους μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ανα μεταξύ των νέων στις διάφορες χώρες και στις διάφορες περιφέρειες υπάρχουν τελείως διαφορετικά επίπεδα γνώσης και ικανοτήτων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Και τώρα εξ ονόμαστε των Σοσιαλιστών, για τρία λεπτά η κυρία Νεντελάτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, χαίρομαι που συζητάμε το Εράσμους. Είναι, ζητώ συγγνώμη που το αποκαλώ έτσι. Ευχαριστώ του συναδέλφου στο Κοινοβούλιο που συνέβαλαν στο να καταλήξουμε σε αυτό το καταπληκτικό κείμενο που ικανοποιεί όλους τους βουλευτές. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Πάγια Τσάοκνες προσπάθειες που έκανε υπέρ των ε, μαθητών, ε, φοιτητών και σπουδαστών. Να συγχαρώ τη Τζούντι Κορέλα και άλλα μέλη της Επιτροπής καθώς και το επιτελείο της κυρίας Βασιλείου. Να ευχαριστήσω επίσης τη Λιθουανική Προεδρία καθώς και την Τζούλια Άντερσον που βοήθησε το Κοινοβούλιο να συντάξει το κείμενο που κατά τη γνώμη μου μπορεί να γίνει αποδεκτό από όλους. Πιστεύω ότι καλύπτονται οι προσδοκίες του Κοινοβουλίου και της επιτροπή μας με το κείμενο. Είναι ξεκάθαρη η δομή του, είναι εύληπτο και Επί της ουσίας θα έλεγα ότι ε, το Λεωνάρντο Ταβίντσι, το Κομένιους, ε, το Γκρούνφιχ, ε, το Εράσμος θα παραμείνουν ως ονόματα. Ο στόχος είναι η πρώτη κινητικότητα των νέων, η διαβίου μάθηση. Διευρύνεται όμως και το πεδίο της συνεργασίας καλύπτοντας την κοινοτομία και την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Την επόμενη επταετία, χάρη στο πρόγραμμα, πάνω από 4 εκατομμύρια νέοι θα μπορέσουν να λάβουν υποτροφίες Όπως και η κυρία Στριγλεύσκα, θα ήθελα να τονίσω ότι 3 εκατομμύρια μαθητές έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτό Ο στόχος ε, βεβαίως ε, δεν είναι ε, μόνο οι νέοι, οι φοιτητέ και οι σπουδαστέ, αλλά και οι ακαδημαϊκοί. Υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την νεολαία επίση, που δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ξεχωριστό προπολογισμό για την κινητικότητα των νέων, για τις οργανώσεις των νέων, για τον εθελοντισμό, για, το, για δράσεις ενεργού πολίτη και ούτω καθεξής. Ε, νέοι από ε, μειονεκτικά κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα δεν πρέπει ε, να ε, αποκλείονται από τα προγράμματα ε, και επίσης να τονίσω ότι ο μηχανισμός εγγύησης ε, των δανείων δεν πρέπει να υποκαταστήσει τις υποτροφίες. Κλείνοντας, να συγχαρώ και τα τρία θεσμικά όργανα για την αγαστή συνεργασία τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος τώρα των φιλελευθέρων, ο κύριος Λόκεγαρ. Βασίλειο, Κύριε Βασιλείου, κύριε Επίτροπε. Κύριε Πακ, θέλω να σας συγχαρώ και τις δύο ονόματος των για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και μια πολύ καλή μεταρρύθμιση. Λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό για τα επόμενα έτη και βλέποντας τα προγράμματα ξεχωριστά, διαπιστώνουμε ότι το Erasmus Plus είναι ένα από τα προγράμματα που είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία στο πλαίσιο του επταετούς ε, μελλοντικού πολυ, πολυετούς πλαισίου. Βέβαια μπορούμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα για το Erasmus Plus. Ποιο, ποια συνέχεια θα δοθεί στο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων διαπίστωσα ότι συχνά τέθηκε το ερώτημα της ποιότητας των προγραμμάτων για τους νέους που πηγαίνουν στο εξωτερικό παίξαμε τα νούμερα, χάρη στις συζητήσεις είχαμε διπλασιασμό του προπολογισμού. Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι τι θα αντλήσουν από την εμπειρία αυτή οι νέοι. Θα βελτιωθεί ή, ή θα βελτιωθούν οι ικανότητές τους. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τις συνθήκες της μετακίνησής τους ε, όταν προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των προγραμμάτων. Εκ νέου, τόσο εξ ονόματος των φιλελευθέρων, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες νίκες και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ξανά στον Πρασίγαν η κυρία Μπεναράμπα του, παρακαλώ. Chers collègues, Συνάδελφοι Επίτροποι, 13,1 ε, δις είναι ο για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή ε, αύξηση 40% σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Οι πράσινοι φυσικά ε, χαίρονται ιδιαίτερα για την άφηση. Με την κρίση που βιώνουμε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να ανταποκρίνει τις προσδοκίες των πολιτών. Γι' αυτό χρειαζόμαστε διπρόσθετες δυνατότητες για την εκπαίδευση και για την κατάρτιση. Ε, αυτά τα προγράμματα υπέρ των μειονεκτούσων ομάδων και κυρίως υπέρ των νέων έχουν ιδιαίτερη σημασία. Όντως θα επενδύσουμε στην νεολαία. Κάθε ευρώ που επενδύουμε σε αυτές τις δράσεις έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση της Ευρώπης καθώς και για το μέλλον της οικονομίας της. Θα ήθελα να τονίσω τρία ζητήματα που δημιουργούν κάποια ερωτηματικά. Πρώτον, ε, δεν μπορούσαμε να καλύψουμε ε, και τους νέους ανέργους ε, στα προγράμματα δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι οι περιφέρειες θα χρησιμοποιήσουν εις το έπακρον την αρχή της επικορικότητας που προβλέπεται στο Εράσμους ΣΥΝ. Τα κράτη-μέλη ποια θέση θα δώσουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στα επιχειρησιακά τους προγράμματα αναρωτιόμαστε. Παρακαλούμε, Επίτροπε, όταν ε, εξετάσετε τα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα ε, των κρατών μελών να μεριμνήσετε ώστε αυτή η πληθυσμιακή ομάδα να είναι στον πυρήνα ε, του προγράμματος ε, διότι δεν, ε, αυτή η ομάδα των νέων δεν μπορεί να λάβει υποτροφία βάση από κονδύλια του ΕΚΤ, παραδείγματο χάρη. Δεύτερον, για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, στο κεφάλαιο 4 του προεκλογισμού της Ένωσης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη το κονδύλι τα προγράμματα συνεργασίας με τις μεσογειακές χώρες θα πρέπει να ενισχυθούν στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Στέφαν Φίλε και με το Συμβούλιο ελπίζουμε να φροντίσετε το ώστε να ε, συναυθεί μια συμφωνία για αυτό το ζήτημα. Τρίτον, ξέρετε ότι εδώ στο Κοινοβούλιο καταφέραμε να θέσουμε ανώτερο όριο για το μηχανισμό εγγύηση ε, των φοιτητικών δανείων ε, για τα μεταπτυχιακά του Εράσμους ΣΥΝ. Ωραία, αλλά δεν είναι αυτό που θα εγγύθει ένα καλύτερο μέλλον για την νεολαία. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής εξέτασης και ελπίζουμε να αναλυθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να τηρούνται κατά γράμμα οι διατάξεις για το μηχανισμό εγγύηση αυτών των δανείων. Η κυρία Μακλάρκιν τώρα από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σίγουρα δόθηκε πολλή δουλειά για την αναδιοργάνωση του προγράμματος αυτού τους τελευταίους 18 μήνες. Και πρέπει να πω ότι ένα χρόνο πριν καταψήφισα την θέση του Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα αυτό. Και η ομάδα μου είχε σοβαρές ανησυχίες για μια σειρά θεμάτων. Το μέγεθος του προπολογισμού και τις μικρές εγγύησεις. Ωστόσο, μετά τους τριλόγους υπό την Ιρλανδική Προεδρία, το κείμενο βελτιώθηκε προς το βελτίο. Δεν είναι το καλύτερο, είναι καλύτερο. Το Εράσμο στη χώρα μου θεωρείται ως κάτι από τα λίγα που δουλεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν προστιθέμενη αξία και ελπίζω το πρόγραμμα αυτό να συνεχιστεί για να μπορέσουν οι νέοι να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες να, μελε... να σπουδάσουν εκτός της χώρας τους μαθαίνοντας από διάφορες κουλτούρες. Ωστόσο, έχω απογοητευθεί και έχω σοβαρές επιφυλάξεις για τα τεράστια ποσά που δίδονται στην χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων Ζαν Μονέ που προωθεί την ευρωπαϊκή ενοποίηση και που καταρτίζει την ελίτ των Βρυξελών. Είναι απαράδεκτο να δαπανά το Κοινοβούλιο περισσότερα κονδύλια για την εκπαίδευση των δικών του γραφειοκρατών από ό,τι για τον αθλητισμό. Τα θετικά τώρα. Για πρώτη φορά ο αθλητισμός πήρε συγκεκριμένο ε, προϋπολογισμό και θα ήθελα να, να λάβει ο αθλητισμός μεγαλύτερο κομμάτι στο εράσμος... αλλά καλωσορίζω διότι την έμφαση στον αθλητισμό της βάσης. Αυτοί θα κερδίσουν περισσότερο από αυτά. Όπως είπα το κείμενο δεν είναι τέλειο, αλλά θα υπερψηφιστεί από την ομάδα μου και εμένα ε, σαν μια ευκαιρία για τους νέους και για την επαγγελματική τους κατάρτιση. Ελπίζω αυτό να βοηθήσει όσους θα μετάσχουν κατόπιν στην ε, βοήθεια για την ευρύτερη οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματο τη Ενωτική Αριστερά το λόγο έχει η κυρία Βερζιά. Παρακαλώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα δημοσιονομικά τωρινά πλαίσια, ε, ε, όσοι παίρνουν υποτροφία από το έρασμο ε, ΣΥΝ θεωρούν ότι έχει γίνει θαύμα. Ξέφυγε και από τις περικοπές του Συμβουλίου και είναι ένα από τα σπάνια προγράμματα που θα έχει σημαντική αύξηση στο τωρινό πολιετές πλαίσιο και χαιρόμαστε φυσικά γιατί οι νέοι είναι βασικοί δικαιούχοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σπάνια υπάρχει τέτοια συνένεση. Παρ' όλα αυτά εμεί θα το καταψηφίσουμε το πρόγραμμα διότι ε, είναι κάζος μπέλη για μας ε, αυτό το θέμα του μηχανισμού εγγύηση των φοιτητικών δανείων. Αντί να τονώνουμε τι υποτροφίε, τι θα ενθαρρύνουμε του φοιτητέ να χρεώνονται για να πληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτοί που είναι στη μειονεκτικότερη θέση είναι αυτοί που δυσκολεύονται να βγουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τι είναι αυτό πάλι. Πάλι ο νεοφιλελευθερισμό Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσουμε αυτό το αμερικανικό σύστημα. Μόνο όσοι έχουν λεφτά θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Ε, όχι, δεν θα αφήσουμε να εκτροχιαστεί έτσι η κατάσταση. Εμεί θέλουμε το πανεπιστήμιο για όλου. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριο Φοντάνα, εξ τη ομάδα του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ καταρχά την εισηγήτρια που είναι και πρόεδρο του Επιτροπή Πολιτισμού, όπου μετέχω, την κυρία Πακ, για τη δουλειά που έκανε και αυτή και όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων, οι ηγητές, γιατί πρέπει να σα πω ότι και εγώ πριν από ένα χρόνο δεν θα είχα πιστέψει ότι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τον προπολογισμό του. Ωστόσο έχουμε μπροστά μας μια αύξηση κατά 14 δισεκατομμύρια ευρώ, 40% ε, σαν ποσοστό για τους νέους που πλήττονται ιδίω από την κρίση αυτή. Άρα είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το Εράσμους είναι ένα από τα προγράμματα εκείνα που είναι μεταξύ των πιο γνωστών στην Ευρώπη και ένα από τα προγράμματα που επιτρέπει στους νέους μας να αυξήσουν τα προσόντα τους και από φοιτητική άποψη αλλά και στην εργασιακή εμπειρία τους. Η σύνδεση μάλιστα που θα δημιουργηθεί μεταξύ του πανεπιστημιακού του ακαδημαϊκού χώρου και, επαγγελμα... και του επαγγελματό είναι ακριβώς κάτι που πρέπει να πετύχουμε στην Ευρώπη και μέσω του προγράμματο αυτού δουλεύουμε για να βελτιώσουμε ακριβώς το μέλλον για τους νέους μας. Θα, θα ευχόμουν λοιπόν να αποτελέσει, να συνεχίσει να αποτελεί αυτό το πρόγραμμα έναν φάρο για, το, για την Ευρώπη και ότι να πείσουμε τους νέους μας ότι δεν είναι μόνο εκδρομή αλλά να υπάρχει και ένας αυστηρότερος έλεγχος των δραστηριοτήτων τους. Πάντως αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπρο και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιβο Μπελέτ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι δύσκολο το οικονομικό πλαίσιο και περίπου θαύμα το γεγονός ότι καταφέραμε να αυξήσουμε ε, τα μέσα και τους πόρους για ε, τον έρασμο. Συγχαρητήρια και στην κυρία Βασιλείου, την κυρία Επίτροπο, αλλά και την κυρία Πακ, που δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλος της. Είναι προφανές ότι τα προγράμματα αυτά είναι εκ των όνου για το μέλλον της Ευρώπης. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Η συνεργασία φοιτητών και εκπαιδευτικών ε, διασυνοριακά είναι από τα καλύτερα ε, όπλα μας απέναντι στο λαϊκισμό και ε, υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για το 2020 θα έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των διασυνοριακά κινούμενων και φοιτητών και εκπαιδευτικών και πραγματικά είναι ε, ε, πολύ σημαντικό ε, να το δούμε ως επένδυση στο μέλλον και να μην γίνουν περικοπές ε, στον προπολογισμό του Εράσμου. Είναι και προς το συμφέρον των κρατών μελών να δίνουν στους φοιτητές και τους μαθητές ε, αυτές τις ευκαιρίες. Το είπε και η κυρία Πακ και η κυρία Μακλάρκιν. Τελικά... Το πρόγραμμα αυτό θέτει και τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. Δεν χρειάζεται η Ευρώπη να ρυθμίζει τον αθλητισμό, το αντίθετο. Αλλά υπάρχουν ε, διάφορα ε, ζητήματα. Κυρία Επίτροπε, τα γνωρίζετε κι εσείς, κατά πολέμηση των στιμένων αγώνων και το ε, ντόπινγκ είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί πανευρωπαϊκά και έχει και προστιθέμενη αξία έτσι αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Κάμερβερτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά για αυτό το θέμα, αλλά ε, επιτέλους καταφέραμε ε, να ξαναφέρουμε ε, στα πόδια του το πρόγραμμα Εράσμους που είχε ανατραπεί. Ε, ταυτόχρονα ξεκαθαρίζουμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι φοιτητές αλλά και οι μαθητές και οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι αλλά και η εξωσχολική εκπαίδευση και μόρφωση. Και να μην ξεχάσω και τον αθλητισμό εδώ. Ε, η μόρφωση και η παιδεία είναι αυταξία, δεν είναι οικονομικό μέγεθος και αγαθό. Ε, γι' αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, να κοιτάξουμε την εργασία των νέων να υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με ξεχωριστή πρικοδότηση για την εργασία των νέων και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης και τα μεμονωμένα προγράμματα Λεωνάρδο Γκρούντβιχ και Κομένιους που είναι επιτυχή θα διατηρήσουν και το όνομά τους και τη φήμη τους και την αναγνωρισιμότητά τους. Με την πρόταση αυτή νομίζω βρήκαμε μια καλή ισορροπία. 11 μεμονωμένα και υποπρογράμματα έχουν ε, ολοκληρωθεί ε, συνενωθεί σε ένα πρόγραμμα για τη μόρφωση, τη μετακίνηση των νέων και επιτέλους τον αθλητισμό. Για πρώτη φορά αναγνωρίζουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τον αθλητισμό και έχουμε κάποιο ελάχιστο περιθώριο ελιγμών εκεί ευρωπαϊκά. Με αυτό το πρόγραμμα, με πάρα πολύ λίγα χρήματα, επιτυχάνουμε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα προώθησης και πραγματικά μπορούμε έτσι να σφυριλατήσουμε ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ε, με το πρόγραμμα αυτό ε, που θα ε, ζουν την Ευρώπη κάθε χρόνο στο πετσί τους χιλιάδες νέοι και αξίζει πραγματικά ε, μεγαλύτερη αναγνώριση και περισσότερα χρήματα. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ της νέας διευκόλυνσης για τους φοιτητές. Γνωρίζω ότι γίνεται πάρα πολύ επικριτικά η συζήτηση, αλλά είναι μια δυνατότητα που αν μη τι άλλο καλό θα ήταν να τη δοκιμάσουμε. Ε, να δίνουμε την ευκαιρία σε περισσότερους φοιτητές να πηγαίνουν για όλες τις σπουδέ στο εξωτερικό και μετά από δυόμιση χρόνια θα δούμε αν οι προσδοκίες μας έχουν επιβεβαιωθεί. Θα ακούσουμε και τις κριτικές φωνές, αλλά αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Σάκε, παρακαλώ. Σχάκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, επειδή συνέδελφοι, οι διεθνεί δεξιότητε για όσου ακολουθούν ακαδημαϊκή ή εκπαιδευτική κατάρτιση βοηθούν ούτω ώστε να εισέλθουν σε μια διεθνοποιημένη αγορά εργασία και δίνονται και λύσει για τα ανεργία των νέων. Όμω, στο Erasmus Σύνε ο φοιτητή πρέπει να είναι στο κέντρο. Λόγω των περικοπών, βλέπουμε ότι το τίμημα είναι υπερβολικά βαρύ για του νέου ε, εξαιτία ε, τη ε, κοινωνικονομική κρίση στην Ευρώπη. Χρειάζεται καλύτερη απόδοση για τι επενδύσει μα. ολοκλήρωση των διαδικασιών και επίση συμπερίληψη των βασικών στοιχείων. Αυτό επιδίωξε το Κοινοβούλιο, ώστε να αποφύγουμε τα μακροσκελή ευχολόγια που θα αποδυναμώσουν τι τελικέ επιδόσει του Εράσμου ΣΥΝ. Αυτό έγινε τώρα. Θα πρέπει όμω για τα 4 εκατομμύρια των δικαιούχων να ασχοληθούμε με την ποιότητα. Ε, με αυτόν τον μηχανισμό ε, για την εγγύηση των δανείων ευελπιστούμε ότι θα αυξηθεί ε, αυτός ο αριθμός. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ποσοστό παραμένει μικρό, είναι 1,5% το συνολικό κονδύλι ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην γυρίσουμε την πλάτη στους νέους που περιμένουν πραγματική πολιτική ηγεσία. Σας ευχαριστούμε κυρία Τρίπελ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε κυρία επίτροπε, Μάλιστα, το πρόγραμμα Εράσμους είναι μια γνήσια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας. Μέχρι τώρα έχουν συμμετάσχει 3 εκατομμύρια φοιτητές. Είναι πραγματικά Πολύ ωραία προσπάθεια και μόνο πέρσι ήταν 50.000. Είναι χαρμόσυνη αυτή η αριθμή. Και καλό είναι που καταφέραμε εμεί ω Κοινοβούλιο στο πρόγραμμα αυτό να διατρανώσουμε ποια είναι τα υποπρογράμματα. Εράσμου, Εράσμου Μούντου, ε, Γκρούντβικ, Λεωνάρδο και Νεολαία σε δράση. Είναι πολύ σημαντικό τα προγράμματα αυτά να παραμείνουν αναγνωρίσιμα. Παρ' όλα αυτά και σήμερα ε, λόγω της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη θα πρέπει να πούμε ότι θα ήταν καλύτερο να δώσουμε κάτι περισσότερο για το Λεωνάρδο. Πρέπει να το πω αυτό λίγο και κάνοντας την αυτοκριτική μας. Και θυμίζω ότι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει πολύ υψηλότερο προεπολογισμό. Υπάρχει με ένα αύξηση αλλά δεν είναι τόσο τεράστια όσο θα έπρεπε για την ε, πολιτική, ε, την ευρωπαϊκή της παιδείας θα ήταν οπωσδήποτε επιθυμητό περισσότεροι νέοι και περισσότεροι σπουδαστέ και φοιτητέ να συμμετέχουν και να είναι και πιο ψηλέ οι υποτροφίε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρο. Και τώρα η <coughs> κυρία Τόμασιτ. Πρόεδρε, εκτιμούμε τι ε, προτάσει τη ηγήτρια για ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα Πάντως η, το αίτημα της για ποιότητα για όλους είναι καθοριστική σημασία για το μελλοντικό πλαίσιο του Εράσμου, ούτω ώστε να παράσχουμε σε όλους την Ευρώπη ανεξάρτητα ηλικία, προσόντων ή ε, εκπαιδευτικής ικανότητας τις ίδιες ευκαιρίες περαιτέρω εκπαίδευση τις θέση τη ηγεσία, για ένα διοικητικό πλαίσιο το πρόγραμμα αυτό σε κάθε κράτος μέλο, όπου βάσει της αρχής της επικουρικότητα τα κράτη-μέλη θα έχουν αρκετή ελευθερία. Εγώ τόνισα ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω την κινητικότητα στην απασχόληση που καταδικάζει τα λιγότερα προηγμένα, εξελιγμένα κράτη. Η κινητικότητα στην εκπαίδευση είναι καλύτερη λύση γιατί επιτρέπει καλύτερη και γρηγότερη κατάρτιση των νέων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Άγνου, παρακαλώ. Well, I won't be congratulating anybody, uh, chairman, what... Δεν νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε κανέναν είναι το Εράσμος, το έχουμε θεοποιήσει αυτό το πρόγραμμα ανταλλαγή. Ε, θα το κάναμε και χωρί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, στα Βρετανικά πανεπιστήμια έχουμε πολύ άριθμα τέτοια προγράμματα και δεν χρειάζεται να είμαστε σε καμία πολιτική ένωση. Το Εράσμο δεν έχει καμία σχέση με την αριστεία στη μάθηση και με κοινικό τρόπο εκμεταλλεύεστε του νέου ε, για να εξυπηρετήσετε πολιτικού ε, σκοπού. Ε, οι τροπολογίε 38 και 42 τι λένε, ότι χρησιμοποιείτε το Εράσμο για την υποστήριξη εξωτερική δράση και προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών καταπληκτικό. θέλετε να φτιάξετε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα με τον αθλητισμό και την ημέρα του αθλητισμού και θα τα βάλουμε όλα στα μπλουζάκια ε, και έτσι θα δίνονται και πολύ ευκολότερα οι θεωρήσει για να προωθηθεί η κινητικότητα. Τι εννοείται, να ανοίξουμε την πόρτα και να μπαίνουν όλοι οι μετανάστε και έρχονται όλοι οι βουλευτέ και το υποστηρίζουν. Μα είπατε ότι είναι αύξηση 40% οι νέοι που έχουν περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ε, και ε, ουσιαστικά ε, αυτό μας κοστίζει 17,2 δις. θέλετε να απαντήσετε σε μια μπλε κάρτα της κυρίας Μαγκίνες, κύριε Άγνιο, υποθέτω, ναι. Παρακαλώ παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, δεν ξέρω αν πρέπει να πω και στον κόπο να του κάνω την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι καμιά φορά ε, ε τηρούμε παθητική στάση και ε, δεν σχολιάζουμε αυτά που λέγονται, αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Σέβεστε καθόλου τους νέους, κύριε Άγνιου, και σέβεστε την ικανότητα που έχουν να διακρίνουν μεταξύ του καλού και του κακού και τη, σέβεστε την δυνατότητα που πρέπει να τους δοθεί να ε, μαθαίνουν και να ζουν αξιοπρεπώς. Ε, τι έχετε να πείτε. Έχω τρεις ε, γιους απάντηση. Δύο είναι στο πανεπιστήμιο, ένας δουλεύει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή, χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους πούν, ε, ε, να τους πει πώς, ε, πόσο σκληρά πρέπει να εργάζονται. Εγώ αυτό είπα ότι εκμεταλλευόμαστε τους νέους, δεν είναι ότι δεν τους σέβομαι, τους εκμεταλλευόμαστε για να ρίχνουμε λεφτά μέσα σε αυτό το πηγάδι και να εξυπηρετούν τους δικούς τους σκοπούς. Εγώ αυτό είπα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σβέρ. Επίτροπε, καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Πάκα για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Χωρίς τις προσπάθειές της, σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχε πετύχει αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Ακόμα, σε εποχή λιτότητας αυξήσαμε το κονδύλι για το Εράσμους κατά 40%. Να συγχαρούμε λοιπόν και τους εαυτούς μας και την Επιτροπή. Είμαι εισηγητής για την έκθεση, ήμουν εισηγητής για το, το 2011 για την έκθεση για τους νέους και την κινητικότητα και είχαμε υπογραμμίσει πόσο σημαντικό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα να εξυπηρετεί τους νέους μεν αλλά και την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε κάνει μια νέα, είχαμε μια νέα ανάλυση και προβληματική της εκπαίδευσης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αφενός εκατομμύρια νέων χωρίς δουλειά και αφετέρου εκατομμύρια θέσεων κενές που δεν μπορούμε να καλύψουμε γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα προσόντα. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε το σύστημα εκπαίδευσης. Αυτό είναι προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία. Εύχομαι εκ νέου συμπερασματικά να τεθεί το νέο πρόγραμμα σε ισχύ ήδη από το 2014. Όσο νωρίτερα ξεκινήσει, τόσο καλύτερα θα εξυπηρετήσει τους πολίτες ε, της ε, Ένωσης, ιδίως τους νέους πολίτες. Ευχαριστούμε. Ο Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκερέρο Σαλόν, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, δύο θέματα ενδιαφέρουν τους νέους. Το ένα είναι αυτό το ζωτικό έργο και θέμα της απασχόλησης. Το δεύτερο δε, η επιθυμία τους να μετέχουν σε μια κοινωνική και πολιτική ενότητα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε εδώ πολύ για την παροχή εκπαίδευσης στους νέους. Μπράβο μας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να μιλούμε και για αυτές τις κοινέ αξίες που το πρόγραμμα Εράσμους επέτρεψε να έχουν. Δηλαδή το ότι πολλοί νέοι αισθάνονται κομμάτι όχι μόνο της πατρίδας τους αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό το ότι αυξάνεται ο προπολογισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιε χώρε, μεταξύ των οποίων και η δική μου η Ισπανία, όπου η μετακίνηση φοιτητών από και προ είναι από τις μεγαλύτερε στην Ευρώπη, δημιούργησε η κυβέρνηση, λέω, αβεβαιότητα για το μέλλον του προγράμματο ενώ θα έπρεπε η κυβέρνηση να το ενισχύσει όσο περισσότερο γινόταν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Μπίνευ, παρακαλώ. Πρόεδρε, μια και είναι εδώ η κυρία Βασιλείου, θέλω να της πω ένα πρόβλημα που έχουμε. Ως πρώην αθλητής, εγώ υποστήριξα τη συμπερίληψη του αθλητισμού στο Εράσμος. Η χρηματοδότηση επιτρέπει σε νέους να δουλέψουν. Το χρήμα όμως δεν είναι το πάνημα. Το κίνητρο έρχεται όταν σου δίνεται η ευκαιρία να μετάσχεις σε, μία, σε έναν αγώνα και να κερδίσεις. Όμως η ευρωπαϊκή και η, ευρωπαϊκή ρυθμική υφίσταται διάκριση ε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα υπάρξουν μόνο έξι ensemble και η ήπειρος υποδοχής θα έχει δύο. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν ε, άλλοι λόγοι για τον αποκλεισμό ευρωπαϊκών χωρών δεδομένης ε, της παρούσης, διαδικασίας, της παρούσης κατάστασης θα βελτιωθεί ε, η παρουσία κάποιων μόνο χωρών εκτός Ευρώπης, της Ρωσίας, του Καζακστάν. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών εις δύο ΔΕ της ρυθμικής. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάντεν Καμπ. Ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, τα πιο προβεβλημένα και τα πιο ορατά για την νεολαία μας και πρέπει να είμαστε περήφανοι και μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα σε καιρούς που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί ε, νέα νομιμότητα και νομίζω ότι οφείλουμε μεγάλες ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στην Doris Πακ που έχει κάνει τεράστια δουλειά ως εισηγήτρια ε, σε αυτό το θέμα που ήταν και περίπλοκο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη διεύρυνση των ομάδων στόχων και ιδιαίτερα στη μέση εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση δηλαδή. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι ότι ε, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι φοιτητές σε θετικές σπουδές ε, αξιοποιούν καλά το Εράσμο. Τώρα όμως ε, πάμε και στην επαγγελματική κατάρτιση και τη δευτεροβάθμια και τους ε, ανθρώπους με αναπηρία και τον αθλητισμό. Και μην μου πείτε ότι δεν είναι εργασία ο αθλητισμός γιατί είναι εκατοντάδες και χιλιάδες οι νέοι που εργάζονται στον αθλητισμό. Και θέλω να πω δύο λόγια για την ανεργία των νέων. Έχω καμιά φορά την εντύπωση ότι ο έρασμος ε, θεωρείται ε, ένα πρόγραμμα γενικό και αόριστο που έχει να κάνει με τις σπουδέ και δεν είναι πολύ καλά προσανατολισμένο στην αγορά εργασίας. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει αυτό να ενισχυθεί. Αν το κάνουμε σήμερα θα έχουμε ε, κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κύριο Σίβαν, παρακαλώ. ένα λεπτό vorbim uh, Ευχαριστώ. Συχνά τα τελευταία χρόνια μιλάμε για την ε, οικονομία χωρίς αποκλεισμού, την ε, διατηρήσιμη και ευφυή οικονομία, την καταπολέμηση της ανεργίας. Και να λοιπόν επιτέλους έχουμε ένα πρόγραμμα στη διάθεσή μας ε, που έχει κλείσει 25 χρόνια λειτουργίας αλλά πλέον τώρα έχει επαναπροσδιοριστεί επακριβέστερα και διαθέτει και αυξημένη χρηματοδότηση. Δεν νοείται ενιαία οικονομία δίχως ενιαία αγορά εργασίας εάν δεν κατοχυρώσουμε την κινητικότητα των νέων, την ανταλλαγή φοιτητών ανάμεσα στα πανεπιστήμια, εάν δεν εξασφαλίσουμε την κινητικότητα των εργαζομένων που θα έχουν φάμιλες δεξιότητες, δεν μπορούμε να μην εξασφαλίσουμε ότι θα είναι όλοι σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καλά προετοιμασμένοι για ε, την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Ε, συγχαίρουμε και την Επιτροπή Προπολογισμών για τη στάση που για την χρηματοδότηση του προγράμματος. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σάντσες Σμιτ τώρα. Merci, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Εράσμος είναι κατά πάσα πιθανότητα το πιο γνωστό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ήταν μεγάλη πρόκληση η ανανέωσή του. Έγινε αυτό τώρα με το Εράσμος ΣΥΝ, χάρη στη δουλειά της Ντόρις Πάκα του Κοινοβουλίου και έχουμε ένα πραγματικό έρισμα για την ε, σύσφυξη των δεσμών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την περίοδο 2014-2020 επιτύχαμε αύξηση 40%. Μεγάλη επιτυχία που καταδεικνύει και τη δέσμευσή μας ε, στον τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης νεολαίας και του αθλητισμού. Με τη δυσχερή, με τη δυσχερή οικονομική συγκυρία που γνωρίζουμε όλοι είναι μεγάλη πρόκληση για τους μέλους. Η διαβίου μάθηση δεν θα μας βοηθήσει να εξέλθουμε από την κρίση και θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε ευφύ διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα απτό πρόγραμμα. Αυτό περιμένουν από εμά οι πολίτες. Έτσι θα αναστρέψουμε το αρνητικό κλίμα και την ευθύνουσα υποστήριξη των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σενάλοβα, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, η εκπαίδευση είναι κλειδί για την ευημερία της Ένωσης στο μέλλον και υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητά μας. Η εκπαίδευση είναι και τυπική και άτυπη. Η κατανόηση των διαφορών χωρών των λαών τους και της κουλτούρας είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσει τα εμπόδια μεταξύ των λαών. Πρέπει να δούμε ένα τον άλλο με τα δικά μας μάτια. Και το Εράσμους είναι η ναυαρχίδα της Ένωσης. Καλωσορίζω την αύξηση του προϋπολογισμού που δείχνει τη σημασία του προγράμματος και επιτρέπει σε 4 εκατομμύρια Ευρωπαίων να κερδίσουν υποτροφίες τα επόμενα έτη. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές, αλλά και εσάς για το αποτέλεσμα. Εξαιρετική δουλειά, μπράβο σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Μπασέσκου, παρακαλώ. Πρόεδρε, θέλω και εγώ να συγχαρώ την κυρία Πακ για την συμβολή της, για την βελτίωση του προγράμματος. Εκτιμώ ιδιαίτερα την έκθεση αυτή, διότι για πρώτη φορά όλα τα προγράμματα του εκπαιδευτικού τομέα συνεργάζονται, εντάσσονται σε ένα νέο πλαίσιο. Πάνω από 14 δις για το πρόγραμμα αυτό. Ένα μήνυμα για την υποστήριξη της Ευρώπης στην εκπαίδευση. Ιδίως να σκεφτούμε την εξαιρετικά υψηλή ενεργία μεταξύ των νέων. Τα κέρδη από το Εράσμους δεν περιορίζονται στην παραμονή ενός φοιτητή σε μια άλλη χώρα. Η παραμονή αυτή διευκολύνει την επαγγελματική κινητικότητα, ε, νέες ιδέες επιχειρηματικότητας στη χώρα προέλευση. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην κινητικότητα των φοιτητών με τις χώρες της Ανατολής. Τα επόμενα έτη θα πρέπει να δοθούν περισσότερες υποτροφίε σε φοιτητέ από τη Μολδαβία. Ευχαριστώ κυρία Παλιαδέλη παρακαλώ. Ένα λεπτό. Το κείμενο που καλούμαστε να ψηφίσουμε αύριο στην Ολομέλεια είναι ίσως ένα από τα καλύτερα δείγματα συνεργασίας ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς αφού στην τελική του μορφή είναι το αποτέλεσμα ενός έντιμου συμβιβασμού σε τομείς που έμοιαζαν στην αρχή εξεπέραστη. Ενώ το νέο τίτλο που διατήρησε ως brand name το πιο πετυχημένο ίσως ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων ευρωπαίων μαθητών φοιτητών και δασκάλων την αναγνωρισιμότητα των επιμέρους προγραμμάτων τη δίκαιη κατανομή των ανάλογων κονδυλίων την οικονομική υποστήριξη μη επαγγελματικών αθλητικών διοργανώσεων και τέλος την επιτυχή διαπραγμάτευση για το ύψος του προπολογισμού με μια αύξηση 40% ε, παρά εν μέσω οικονομικής κρίσης κρατώ ομολογουμένως τις επιφυλάξεις μου για την αποτελεσματικότητα των φοιτητικών δανείων αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την επίτροπο παιδείας και πολιτισμού κυρία ανδρούλα βασιλείου που θέλησε να νοικοκυρέψει πραγματικά κάτω από την ίδια ομπρέλα διάσπαρτα μέχρι πριν από λίγο καιρό προγράμματα την πρόεδρο της επιτροπής πολιτισμού κυρία Ντόρις Πάκ, για την αγωνιστικότητα και την αγάπη της στους νέους και βεβαίως τους σκιώδεις εισηγητές που συνέβαλαν στην τελική διαμόρφωση του επταετούς προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Μετσόλα. Μια ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την κυρία Πακ για την εξαιρετική δουλειά που έκανε στο θέμα αυτό. Ήμουν από τις πρώτες ερασμίτισες φοιτήτριε και ξέρω από πρώτο χέρι τι ήταν το πρόγραμμα. Ή καταλαβαίνω τη σημασία της πανεπιστημιακής κινητικότητας για να διαμορφωθεί μια ενεργή ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Πρέπει να μπορούμε να επενδύσουμε στους φοιτητές και να επιτρέψουμε στις χώρες να επενδύσουν περισσότερο στην παιδεία για να μπορέσουν οι σημερινοί φοιτητέ να γίνουν οι ηγέτες του αύριο. Με τα προγράμματα κινητικότητας αυτό επιτυγχάνουμε. Εγώ ως Ευρωβουλευτής μπορώ σήμερα πραγματικά να τιμήσω το Εράσμους ψηφίζοντας αυτή την τροπολογία που θα καλύψει και θα αφορά πάνω από 4 εκατομμύρια νέους στην Ευρώπη που θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να μελετήσουν, να δουλέψουν ή να κάνουν θελοντισμό στο εξωτερικό. Ευχαριστώ την κυρία Πάκ, ευχαριστώ την Επίτροπο. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που πετύχανουμε. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Η ε, κυρία Κώστα, γι' αυτο που πετυγχάνουμε. ευχαριστω λεπτό. κυρια ε, κωστα σημαντικό ότι τη χρονιά της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας ξεκινήσαμε για την επόμενη επταετία με μια σημαντική αύξηση του προπολογισμού και πραγματικά μετά από αίτημα και δικό μας και της Επιτροπής το πρόγραμμα Εράσμους που είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής ηθαγένειας για, τους νέ, για τις νέες γενιές μαζί με το Ερκομένιους Λεωνάρντο που επιτρέπουν στους φοιτητές και της ε, δευτεροβάθμιας και της ανώτερης εκπαίδευσης να μετακινηθούν. Μαζί με την εισηγήτρια υποστηρίξαμε τη διατήρηση του Erasmus Plus για την, το, σήμα, βελτιώντας ωστόσο το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για δάνεια και μάστερ, προσωπροθώντας την εμπειρία για την υποστήριξη έργων και δραστηριοτήτων των ε, οργανώσεων νέων και για την υποστήριξη της Ευρώπης στα προγράμματα Ζαν Μονέ με, παράλληλα με ένα ειδικό κονδύλι για τον αθλητισμό. Προσφέρει στους νέους ε, την δυνατότητα και δίνει το μήνυμα ότι η Ευρώπη θέλει να ξαναρχίσει να λειτουργεί από τους νέους. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάτο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Προσφέρουμε λέμε ναι ξεκάθαρα στο πρόγραμμα, εράσμου. πρόγραμμα Ωστόσο δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε τη λύπη μας για την έκφραση της θέσης του, του, του, του Επιτρόπου ε, ε, Παιδί Εκπαίδευσης για τη θέση της κυβέρνησης Ισπανίας. Μην το ξεχάσετε, η Ισπανία ήταν αυτή που μεταξύ των πρώτων συνέβαλε και εγγυάτως τους φοιτητές την δυνατότητα να μετακινηθούν με βάση το πρόγραμμα αυτό. Μην ανησυχείτε λοιπόν. Ε, γι' αυτό. Καλωσορίζουμε το νέο πρόγραμμα που είναι πολύ πιο ξεκάθαρο και επιτρέπει συγχώνευση των διαφόρων ε, ξεχωριστών δραστηριοτήτων ενώ περιλαμβάνει για πρώτη φορά και τον αθλητισμό. Περισσότερο Εράσμους συμπεριμένει περισσότερες ευκαιρίες και γι' αυτό το λόγο είμαι βέβαιος ότι το μέλλον του Εράσμους είναι εξασφαλισμένο. Οι νέοι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι δεν θα επιτρέψουμε κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ο κύριος Στήρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χάρη σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, 5 εκατομμύρια νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν ή να ακολουθήσουν κάποια εκπαιδευτική κατάρτιση στην Αλοδαπή, των οποίων 3 εκατομμύρια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία και έτσι ε, θα ε, πλησιάσουμε την ολοκλήρωση της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μόνο έτσι θα έχουμε συγκριτικό πλενέκτημα στην Ευρώπη λόγω της παγκοσμιοποίησης, αλλαγής των διεθνών σχέσεων και άλλων αναγκών θα πρέπει να ενισχυθεί η διαβίου μάθηση. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση λοιπόν και η εκπαιδευση η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχουν ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Κροατία. 52% των νέων είναι άνεργοι στην Κροατία. Χρειαζόμαστε αυτή την επένδυση είναι η καλύτερη δυνατή επένδυση για το μέλλον της Κροατίας και το μέλλον της νεολαίας στην Κροατία. Κύριε Σκούρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κρίμα πρόεδρε που η συζήτηση αυτή γίνεται μια μέρα που ακόμα πολλοί βουλευτές ταξιδεύουν αλλά και δεν είναι παρόντες πολλοί επισκέπτες γιατί είναι βασικό για το μέλλον της Ένωσης και θέλω να υπογραμμίσω την εξαιρετική δουλειά που έκανε η συγκεκριμένη κυρία Πακ, φτάνει και για χάρη στις ικανότητες της Επιτρόπου κυρίας Βασιλείου να καταλάβει τις απαιτήσει του Κοινοβουλίου. Το Εράσμος, το Λεωνάρντο, το Κομένιους ε, είναι, είναι προγράμματα που φτιάξαν περισσότερο την Ευρώπη από τις ποσοστώσεις του γάλακτος γιατί δεν διέρεσαν, δεν δημιούργησαν ε, διαδηλώσεις κατά των Βρυξελών, αλλά ένωσαν, δημιούργησαν ευαισθησίες, φιλίες, επέτρεψαν στους νέους να γνωρίσουν την Ευρώπη με τις διαφορές αλλά και να δημιουργήσουμε μια κοινή βάση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την εμπειρία αυτή. Ήταν σημαντικό με το Erasmus Plus να προσανατολίσουμε το, ε, το πρόγραμμα προς την κατεύθυνση αυτή. Σήμερα χτίζουμε ένα μικρό κομμάτακι ακόμα Ευρώπης, της πραγματικής Ευρώπης, των νέων, των φοιτητών, όχι των γραφειοκρατών. Φτιάχνουμε μια Ευρώπη που είχαν φανταστεί πριν από πολλά χρόνια οι ιδρυτές της Ευρώπης. Γι' αυτό μπράβο. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι φτάσαμε στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΗ. Πάνω από 26 συνάδελφοι έχουν εγγραφεί, έχουν ζητήσει το λόγο. Αλλά ε, τα μάτια μου δεν βλέπουν τόσο πολλούς, δεν μπορώ να δω 26 συναδέλφους. Μέχρι 8 βλέπω. Μέχρι 8 συναδέλφους μπορώ να αναγνωρίσω. Και αναλογικότητα από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Θα δώσω πρώτο το λόγο στην κυρία Ζαμπόρσκα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε Βασιλείου, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας την κυρία Ντόρι Πακ. Εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά και εντατικά για την ε, μεταρρύθμιση του προγράμματος Εράσμους. Πιστεύω ότι θα επαρκέσουν τα κονδύλια και δεν θα επαναληφθεί η πρόσφατη κρίση που χρειάστηκε να επιλύσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα. Το χρηματοδοτικό εργαλείο, ο μηχανισμός εγγύησης των φοιτητικών δανείων ε, στην Αλοδαπή είναι ένα νέο και σημαντικό στοιχείο, διότι έτσι διευρύνεται το φάσμα των επιλογών των νέων. Το μέλλον της Ευρώπης είναι συνάρτηση της κινητικότητας των νέων της. Έχουμε μια ολόκληρη νέα γενιά που μπορεί να ταξιδέψει και να γνωρίσει από κοντά την υπόλοιπη Ευρώπη, να οικοδομήσει σχέσεις ε, με την υπόλοιπη Ευρώπη και να κατανοήσει για ποιο λόγο ε, είναι λένθα το πεπρωμένο μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Επόμενος, επόμενη, κυρία Γιώψεβα. Господин председател, програмирането на Еразъм за всички е очакваната стъпка към усъвършенстване на механизмите за... Подойде το Εδάσμους για όλους είναι το αναμενόμενο βήμα για τη βελτίωση μηχανισμών συνεργασίας, εκπαίδευσης και αθλητισμού. Ο τελικός στόχος είναι να επιτευχθούν ε, οι στόχοι της Ευρώπης του 2020. Η εκπαίδευση προφανώς είναι τομέας προτεραιότητας. Θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, η υποστήριξη για την καινοτομία θα βελτιώσει την, ε, τα κίνητρα των νέων. Δεύτερον, τα προγράμματα θα είναι επιτυχέστερα αν επανεξετάσουμε τις ε, διαδικασίες απλοποιώντας τις, εναρμονίζοντας για παράδειγμα τις οικονομικές προϋποθέσεις για τις διάφορες δραστηριότητε. Οι, διάφορες, ε, οι διαφορετικοί συντελεστές για φοιτητέ και καθηγητές θέτει κάποιες χώρες σε λιγότερο ευνοϊκή θέση, κάνοντάς τις δηλαδή λιγότερο οικιστικό προορισμό. Η πληρωμή σε άτομα που μετέχουν στην ίδια δομή διαφορετικών υποτροφιών δημιουργεί κακές σχέσεις. Πρέπει να δημιουργήσουμε καλύτερη συνεργασία. Οι διαδικασίες απλοποίησης ελπίζω να επανεξεταστούν γιατί είναι βασική προϋπόθεση επιτυχίας. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Μπιλμπάου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη βελτίωση της πρικοδότησης του προγράμματος «Έρασμος για όλους». Έχει καλύτερη δομή και μεγαλύτερη σαφήνεια για τους ε, δικαιούχους. Θα έχει και περισσότερους πόρους για ε, την επόμενη περίοδο 2014-2020 ε, από τα τρία ε, δις αυξάνεται σημαντικά. Είναι μεγάλο επίτευγμα και δείχνει ότι η Ευρώπη ε, πραγματικά χρησιμεύει σε κάτι. Βελτιώνεται ένα πρόγραμμα που είναι υπέρ των νέων, που τους βοηθάει, τους βοηθάει να κυκλοφορούν στην Ευρώπη και να δημιουργούν γνωριμίες και να, συνδέσεις. πάνω από 4% αυξάνεται ε, στη Μαδρίτη όμως ε, γίνονται περικοπές και στην παιδεία. Δεν θέλει ε, η Ισπανική κυβέρνηση σήμερα να βελτιώσει την ευρωπαϊκή πορεία των φοιτητών της. Θέλει να τους περιορίσει την Ισπανία. Thank um, Ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι ο Εράσμος ε, σε ένα σύγγραμμα του ε, καταγγέλει ε, ε, την, ε, θεο, τους θεολόγους παραδείγματος χάρη πριν από 500 χρόνια και λέει ότι ε, με αυτόν τον κεραυνό θα τρομάξω όσους δεν συμφωνούν μαζί μου. Ε, τι κάνουν, συμπεριφέρονται σαν να είναι ήδη στον παράδεισο και κοιτάζουν με λύπηση τους υπόλοιπους σαν σκουλίκια. Ε, βγάζουν συμπεράσματα, κάνουν υπονοούμενα, ε, ε, είναι πολυλογάδες ε, και βρίσκουν συνέχεια νέους εύσχημους όρους. Νομίζω ότι αυτή την περιγραφή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να χαρακτηρίσουμε το Erasmus In που είναι η μεγαλύτερη τρέλα του δικού μας αιώνα. Ευχαριστούμε ο κύριος Μποργέζιο τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι από την ε, κοινοβουλευτική μάχη που δώσαμε για να αποφύγουμε να εξαφανιστεί το Εράσμους. Με εκπλήσει όμως ε, που άκουσα εδώ πέρα ότι είπαν ότι ο στόχος ήταν λάθος και ότι το Εράσμους ε, εξομαλύνει διαφορές. Εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρατήσει τις διάφορες κουλτούρες. Αν ο στόχος του Εράσμου ήταν να ισοπεδώσει τις διαφορές θα ήταν λάθος. Όχι. Οι προτάσεις που προήρθαν από το, ε, είναι Φερρυπίν η ανταλλαγή κατοικίας με μείωση με αύξηση των ε, δυνατοτήτων ε, δουλειά ε, σε διάφορες χώρες. Το Εράσμους δεν πρέπει να γίνει γραφειοκρατία των Βρυξελών, αλλά να εκφράσει ό,τι καλύτερο υπάρχει από τον πολιτισμό και την συνείδηση της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριος Τσάμπα Σόγουρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμα Εράσμος είναι το πιο γνωστό πρόγραμμα σε όλη την Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτό. Και μάλιστα και το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα είναι για εκατομμύρια φοιτητέ. Δεν είναι μόνο ένα εξάμεινο στο εξωτερικό και νέε γνωριμίες, αλλά ε, γνωρίζει και την Ευρώπη νεολαία και ε, ζει την ευρωπαϊκή ταυτότητα και πραγματικότητα καθημερινά προσαρμόζεται σε νέες προκλήσεις και ψεύεται ο ένας τον άλλον. Η κοινή Ευρώπη λοιπόν δεν ενσαρκώνεται από κανένα πρόγραμμα καλύτερα από, από τον έρασμο ε, γιατί οι νέοι πραγματικά διαμορφώνουν το μέλλον της Υπήρου μας. Καλό είναι που ξεπεράστηκαν τα χρηματοδοτικά εμπόδια και στην επόμενη προγραμματική περίοδο ε, δεν τίθεται ε, τέτοιο θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Νταντζίλα. susțin propunerea comisiei europene și a raportoarei privind modificarea structurii regulamentului ε, με την πρόταση για τροποποίηση της δομής του κανονισμού ώστε να εντοπιστούν καλύτερα τα υποπρογράμματα ανα εκπαίδευση και κατάρτιση επιτυγχάνουμε και καλύτερη οριοθέτηση των στόχων κάθε προγράμματος. Έχουμε επίσης αγωγή ενός νέου προγράμματος για τον εθλητισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, διαφυρώσουμε συγγνώμη, το χάσμα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ε, την ε, διαβίου μάθηση με την αγορά εργασίας για να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης της ανεργίας, κυρίως καταπολέμησης ε, της ανεργίας των νέων, καλύπτοντας πλέον και τον τομέα του αθλητισμού. Υποστηρίζονται πλέον ειδικότερα προγράμματα για άτομα με αναπηρίες ή που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Ε, ε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με, την, ε, με το νέο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε κύριο Στάκουλα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βασίλειο για αυτή την καλή πρωτοβουλία, τη σωστή πρόταση διπλασιάστηκε ο προπολογισμό, μεγάλο, επιτυχή, μεγάλο επίτευγμα. Μπράβο στην κυρία Ντόρι Πακ, πρόεδρο της Επιτροπής μας, έκανε καλή δουλειά, πρωτοπορώντας τον τομέα αυτό. Νομίζω ότι οι δύο κυρίες αυτές έκαναν μια εξαιρετική δουλειά, πολύ καλή για την Ευρώπη. Το Εράσμους θα μεταφέρει τους νέου από τη μια χώρα στην άλλη όπω έκανε στο παρελθόν και πρέπει να επενδύσουμε στους νέου, στην καινοτομία, στην έρευνα, στην κινητικότητα γιατί στην Ευρώπη υπάρχει ύφεση και πρέπει να χτίσουμε μια γέφυρα για το μέλλον. Αυτό κάνει το πρόγραμμα αυτό, αυτό είναι το πρόγραμμα αυτό. Και χαίρομαι που δεν καταλήψαμε και τον αθλητισμό και το συμπεριλάβαμε στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ ο στον ομιλητών στη διαδικασία Κατσιάη. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ε, Just a minute, please. Διακόπτει ο Πρόεδρος, μια στιγμή παρακαλώ. Mr. Migalski. Ο κύριος Μιγάλσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, το Εράσμος είναι ένα από τα προγράμματα εκείνα που περιμένουν οι νέοι στην Ευρώπη με κομμένη την ανάσα και είναι ένα από τα σημαντικότερα νομοθετικά επιτεύγματα της Επιτροπής Εκπαίδευσης με συμφωνία όλων μας σχεδόν που πιστεύουμε ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να επενδύουμε τα χρήματα αυτά. Η πολιτική μου ομάδα μερικές φορές ε, ε εντυπωσιάζεται, αμφισβητεί κάποιες πληρωμές ε, της Ένωσης, αλλά το πρόγραμμα αυτό είναι επένδυση. Επένδυση στους νέους, την εκπαίδευσή τους, στην ικανότητά τους να μάθουν άλλους ανθρώπους, άλλες κουλτούρες, άλλο κόσμο. Αυτό είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον. Ευχαριστώ όλους σας. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ποιος έχει δικαστικό θέμα, η κυρία Μαγκίνες. Ε, πρόεδρε, σύντομο. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά σας. Υπάρχει κανένας γραπτός ή άγραφος κανόνας ότι όταν κάνεις παρέμβαση με ε, μπλε κάρτα δεν μπορείς να πάρεις το λόγο στο Catch the Eye. Ήταν καλή συζήτηση και θέλω να συγχαρώ την Doris Park, ιδιαίτερα για την πολύ σκληρή δουλειά που έκανε και να πω ότι θέλουμε ε, να καταλάβουν οι φοιτητέ ότι είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόεδρε ευχαριστώ και για την ανοχή σας. Ε, δεν υπάρχει γραπτός κανόνας ούτε γραπτός κανόνας όποιος θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει, γιατί εξαρτάται τελείω από τον πρόεδρο. Όποιον δει ο πρόεδρος. Αυτό ε, απαντώ, αλλά πολύ έντεχνα χρησιμοποιήσετε το διαδικαστικό για να ευχαριστήσετε την κυρία Πάκ και να πείτε αυτά που είχατε να πείτε. Και τώρα θα ήθελα να σας θυμίσω, όπως έλεγα προηγουμένως, ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν γραπτός αυτά που δεν μπόρεσαν να πούν εδώ στη διαδικασία του ΚΑΤΣΙΑΙ και θα επισυναυθούν στα πρακτικά. Κυρία Μόρβαη, έχετε διαδικαστικό τώρα. No, blue card is... Γαλάζια κάρτα, τι γαλάζια κάρτα, δεν υπάρχει στο ΚΑΤΣΙΑΙ γαλάζια κάρτα σε αυτή τη φάση της ε, συζήτησης. Παρακαλώ, η κυρία Επίτροπο έχει το λόγο για να ολοκληρώσει από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους αξιότιμους βουλευτές. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον Τόρι Σπά και του σκιώδει εισηγητέ και όλους του υπόλοιπου βουλευτές που συνέβαλαν για τη δέσμευση, την προσήλωση και τη σκληρή δουλειά του. Ω προ την τροποποίηση του ε, κανονισμού Εράσμου. Να τονίσω και πάλι ότι όλοι θα πρέπει να νιώθουμε ικανοποιημένοι χάρη στην ε, ε, αύξηση 40% τη χρηματοδότησης, ενώ σε όλου του υπόλοιπου τομεί περικόπτουν τα κονδύλια. Αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται το πόσο επίγον είναι να βελτιωθεί η πολιτική τη διαβίου μάθησης, εκπαίδευση και τη κατάρτιση των νόεων και αντιλαμβανόμαστε πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα ε, της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης. Είναι λοιπόν ισχυρό το εργαλείο και θα ε, σημάνει μια σημαντική διαφορά στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ε, Ευρωπαίων. Το μικρό κονδύλι του αθλητισμού χαίρομαι που ικανοποίησε πολλούς βουλευτές. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με το κεφάλαιο 4. Είναι ευθύνη και του Κοινοβουλίου για να ψηφιστεί να παρκές κονδύλι για το Εράσμους ΣΥΝΕ στα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ε, εξωτερική δράση. Και απευθύνω έκκληση προς εσά λοιπόν να υποστηρίξετε αυτή την πρόταση. Κυρίες και κύριοι, έχει αναδειχθεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το Εράσμους ε, γιατί συμβολίζει βασικές ευρωπαϊκές αξίες. Ας ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή την υπέροχη ιστορία με το Εράσμους ε, ΣΥΝ για το οποίο μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Ντόρις Πακ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, τέσσερα λεπτά μίλησα προηγουμένω μόνο. Θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά που δεν πρόλαβα να πω. Χαίρομαι που όλοι αγωνιστήκαμε το πρόγραμμα για την νεολαία, η άτυπη μάθηση να συμπεριληφθεί εδώ με ένα ιδιαίτερο προπολογισμό. Ήταν πολύ μεγάλη μου αγωνία και πραγματικά πέρασε. Θέλω να θυμίσω το θέμα του Γκρούντβιχ, που είναι η μετακπαίδευση των ενηλίκων. Είναι σημαντικότερο από ποτέ. Ε, θυμάστε ε, τη μελέτη που λέγει ε, πόσο υπολοιπόμεθα όλες οι χώρες και δεν ξέρω και τη δική μου. Ε, έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ. Θυμίζω ότι στο πρόγραμμα για την νεολαία υπάρχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Εθελοντική Θητεία. Είδα το φθινόπωρο 350 νέους Γερμανούς που πήγαν εθελοντές σηκώθηκε και μου είπε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που ήταν στη Λιθουανία 12 μήνες και τώρα γνωρίζω εγώ τι είμαι, ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Αυτό θέλουμε, έτσι οι νέοι μας να μαθαίνουν ε, πού είναι η θέση τους στην κοινωνία, όχι μόνο αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο, αλλά και αυτά που μαθαίνουν σε ένα διαπολιτισμικό επίπεδο και περιβάλλον. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε σε καλό δρόμο με αυτό το πρόγραμμα και επίση να θυμίσω ότι συμμετέχουν και χώρε εκτό Ένωση, υποψήφιε χώρε. Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν. Το ανοίγουμε για τα κράτη τη Νότια Όχθη Μεσογείου και για την Ανατολική Ευρώπη. Νομίζω ότι με αυτό το πρόγραμμα πραγματικά πήγαμε στο δρόμο που έπρεπε για να είναι καλύτερη η Ευρώπη από αυτές τις ανοησίες που είπαν εκεί απέναντι δύο κύριοι για τον Εράσμο. Κρίμα που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει αμέσως σε αυτές τις ε, ανοησίες. Στο τέλος της συζήτησης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν μαζί μου σε αυτό το θέμα και ε, ε, ιδιαίτερα τους ε, την κυρία Βασιλείου έτσι και αλλιώ, αλλά και τους συνεργάτες σας, ε, κυρία Βασιλείου. Είχαμε μια πάρα πολύ εντατική ανταλλαγή απόψεων. Διαπληκτιστήκαμε κιόλα. Ε, τελικά τα βρήκαμε και αύριο μπορούμε να ψηφίσουμε όλοι το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και πάλι και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο που δυστυχώ απουσιάζει. Ήταν καταπληκτική αυτή η δουλειά και χαίρομαι που στο τέλο των 25 χρόνων θητείας μου κατάφερα να πετύχω αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ ε, με τη σειρά μου, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση, μια σύντομη παρατήρηση να κάνω. Είμαι βέβαιος ότι στον καιρό του Εράσμου επίσης ε, μετακινούνται οι σπουδαστές και οι φοιτητές. Από τότε δεν είναι τίποτα καινούριο. Αλλά αυτοί που ζουν εδώ σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης δεν θα καταλάβουν ίσως ότι για μας που ερχόμαστε από το σιδηρόν παραπέτασμα αυτή η ελευθερία κίνησης ε, τι σπουδαίο σημαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, προσπάθειές σας. Αύριο το μεσημέρι ψηφίζουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπαίνουμε στο επόμενο σημείο της μερικής διάταξης έκθεση της κυρίας Κώστα για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.